Il Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno alla signora commissaria. Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Επίτροπο, στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Καλημέρα σε όλου του αξιότιμου συναδέλφου, άντρες και γυναίκε. Ξεκινάμε τη συζήτησή μα. ξεκινάει η συνεδρίαση. Πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη αφορά την σύσταση τη κυρία Σοφή Ιντβέλτ όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων επιβατών ε, στο Υπουργείο Εσωτερική Ασφαλεία των ΗΠΑ. Τώρα δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, την συνάδελφο κυρία Σοφία Ιντβέλτ, για τέσσερα λεπτά. Έχει λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στον κύριο Επίτροπο. Σήμερα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, αυτή η διαδρομή, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2003. Και για αυτόν τον λόγο έχουμε και αυτήν την υπερατλαντική συμφωνία όσον αφορά την